Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καθίστε σα παρακαλώ πολύ. Να μην ε, αρχίσουμε σήμερα με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Η συγγήτρια κυρία Περβάς ε, Μπερέζ έρχεται. όπου να είναι θα φτάσει. Ε, αξιοποιώ το χρόνο λίγο για να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις και να διεκπαιρεώσουμε μερικά διοικητικά θέματα γρήγορα. Είμαστε πλήρης από διερμηνία σήμερα, έχουμε όλες τις γλώσσες, μπορείτε να μιλήσετε όλη τη μητρική σας γλώσσα. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Κανείς δεν επιθυμεί συμπληρώσει αλλαγές και εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ούτε ανακοινώσει έχω ειδικά σήμερα εγώ. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι... Σήμερα καταθέτει επίσημα υπερβάνς στην έκθεσή της ε, και αύριο θα σταλεί στη μετάφραση, γιατί είναι στα γαλλικά η έκθεση. Γνωρίζετε ότι καταφέραμε να επιβάλλουμε να μεταφραστεί και στα αγγλικά η έκθεση γρήγορα και ε, στις 17 Μαΐου να ε, υπάρχει μεταφρασμένη στα αγγλικά. Αν δεν διαφωνεί η υπερβάνς, που νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει, θα φροντίσω ήδη από αύριο στα γαλλικά ε, να ε, διανεμηθεί η έκθεση. Protokoll vom, unserer letzten Sitzung vom 18. März verteilt. Äh, Σας έχω διανύμει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης 18 Μαρτίου καθώ και τη τελευταία ε, συνάντηση των συντονιστών τη 29 Απριλίου δηλαδή και η σημερινή συνεδρίαση με τη μορφή αυτή τουλάχιστον είναι η τελευταία πριν από τις ε, θερινές διακοπέ. Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας που έχει συντάξει η συνάδελφός μας κυρία Ρεγκίνα Βαστός. οικονομικές στρατηγικές εξόδου, οικονομικές και νομισματικές πτυχές, ΜΜΕ, καινοτομία και νέες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα είναι ευρύ φάσμα θεμάτων, οφείλω να το ομολογήσω, και επίσης οφείλω να εκφράσω την, ε, τον θαυμασμό μου για την εργασία της ε, συναδέλφου μας η οποία μπόρεσε να ε, μελετήσει και να συντάξει την έκθεση αυτή τόσο γρήγορα. Καλώς ήρθατε Περβάνς. Θα παρακαλέσω λοιπόν την ε, ε, Ρεζίνα Μπαστός να αναπτύξει σύντομα βέβαια τις βασικές γραμμές της εκθέσεώς της ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε προβλέψει όπως θα είδατε στην ημερήσια διάταξη χρόνο συζητήσεως μέχρι τις 5 η ώρα χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε το χρονικό αυτό περιθώριο. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο επίσημα στην Ρεζίνα Μπάστος, θα καλωσορίσω μια ομάδα φοιτητών της πρωτοβουλίας Focus Ευρώπης. Όχι μόνο λόγω των ενδιαφερόντων τους, αλλά και λόγω της εξαιρετικής τους απόδοσης. Έχουν προσκληθεί λοιπόν τα πρόσωπα αυτά να επισκεφτούν εδώ τις Βρυξέλλες και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκφράζω τη χαρά μου που οι ε, νέοι οι Ευρωπαίοι νέοι ενδιαφέρονται για την ε, για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω για, την, ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά θα προσέλθει και άλλη ομάδα επισκεπτών από κάπως πιο ηλικιωμένους κυρίους που είτε είναι συνταξιούχοι του ε, οικονομικού ε, τομέα. Η κυρία Ρεζίνα Μπάστος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σήμερα η παρουσίαση της, του θεματικού μου εγγράφου συμπίπτει με την ε, παρουσίαση της έκθεσης της εισηγήτριας Μπερές ε, Περβάος. Ελπίζω πως η συμβολή μου θα είναι χρήσιμη για την εκπόνηση της τελικής έκθεσης και ότι αυτή η δική μου παρουσίαση έχει στόχο να εστιάσει στα θέματα του τίτλου, αλλά και σε μια ιδιαίτερη πτυχή που αφορά την υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν να μπούμε στις βασικές ε, συστάσεις που εκθέτω στο έγγραφο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ολόκληρο το έγγραφό μου διέπεται από αξίες οι οποίες θα πρέπει να μας χαρακτηρίζουν στη σημερινή και μελλοντική φάση με την έξοδο δηλαδή της κρίσης που είναι η ελευθερία, η ελεγγύη και η ευθύνη, η υπευθυνότητα. Θα ήθελα αυτές οι αξίες να συμπεριληφθούν επίσης στην τελική έκθεση και ότι η κοινωνική πτυχή που συνδέεται με τις τρεις σπουδαίες αυτές αξίες θα να επεξηγηθεί ε, σωστά στην έκθεση γιατί η κρίση την οποία διανύουμε, εκτός από χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική, είναι και κρίση αξιών. Περνώ στις συστάσεις, τις οποίες εκθέτω στο θεματικό μου έγγραφο και θα ήθελα να τονίσω πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι γνωστό, αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό και ένα από τα σημαντικά ε, μέτρα για την έξοδο από την κρίση για την ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να είναι το στίχημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις αξίες ε, για ε, την εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτού του αιώνα. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς, την υποστηρίζουμε, αποφεύγοντας τις τάσεις που επικρατούν σε αυτές τις περιόδους ε, για θέμη του ανταγωνισμού. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για την μεγάλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχει σχέση με την ε, ενισχύσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι η βοήθεια που έδωσαν τα κράτη στις τράπεζές τους με, αμέσως μόλις ξέσπασε η μεγάλη οικονομική κρίση ήταν ε, ενισχύσεις οι οποίες προορίζοντας προορίζονταν για τις μικρομεσαίες ε, ε, επιχειρήσεις και αυτές τώρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην πρόσβαση σε πιστώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχουν ε, καθεστώτα που θα εγγυώνται τις πιστώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα έχουμε να ασχοληθούμε και με τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και τις δυνατότητες της νέες ευκαιρίες για ε, εμπόριο που ανοίγονται. Θα πρέπει να αποτελέσουν μια διευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα εξασφαλίσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, την πρόσβαση σε αυτές τις νέες ευκαιρίες που με διαφορετική μορφή δεν θα την είχαν. Αυτή η πλατφόρμα για τις ε, ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελούσε ένα πολύ χρήσιμο μέσο εργαλείο ώστε να δημιουργηθεί ένα γόνιμο κλίμα για το εμπόριο αλλά και για να υπάρξει συμπληρωματικότητα με τις ενέργειες των επιχειρήσεων που μπορεί να είναι διευρωπαϊκές στις ε, δραστηριότητές τους. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τον εμπορικό αυτό τομέα, το Small Business Act, θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που θα το καθιστήσουν, καταστήσουν πιο ε, ευκίνητο και θα διευκολύνουν τη λειτουργία του. Αυτό λοιπόν το Small Business Act θα πρέπει να αναθεωρηθεί και γι' αυτό και ζητώ από την ε, εισηγήτρια που αναφέρεται σε αυτό στην έκθεσή της να μεταρρυθμιστεί ώστε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει μια εποπτεία είναι βέβαια κυρίως ε, ε, ευθύνη των κρατών μελών και θα πρέπει ωστόσο να αποδοθεί σε αυτήν την πράξη μια πιο ευρεία κοινωνική πτυχή. Οι μικρομεσαίες, όπως γνωρίζουμε, δημιουργούν νέε θέσει απασχόλησης και οδηγούν σε μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ένα μέτρο συγκεκριμένο που προτείνουμε, γιατί σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για συγκεκριμένα μέτρα, είναι ένα, μια νέα θηρίδα για όλα τα διοικητικά θέματα που αφορούν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τα γραφειοκρατικά διαχειριστικά θέματα θα πρέπει να διευκολυνθούν, να ξεπεραστούν και αυτή η ενιαία θηρίδα, το η οποία ήδη βλέπουμε να εφαρμόζεται σε κάποια κρατημέλη, χρειάζεται μια νέα όθηση ώστε με τη σειρά τη να παροτρύνει και να εθαρρύνει τον ευρωπαϊκό εμπορικό κόσμο. Μια άλλη πρωτοβουλία που προτείνεται έχει σχέση με την ωφελόμενη εκτίμηση, αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουμε για το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, δηλαδή δηλαδή να δημιουργηθεί μια, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ηλικιωμένων συμβούλων. Τι σημαίνει αυτή η ιδέα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι δημιουργούν περισσότερη προστιθέμενη αξία και που βρίσκονται σε μια τελική φάση του επαγγελματικού τους βίου και που περιμένουν και βλέπουν την φυσιολογική τους απομάκρυνση από την αγορά εργασίας μπορούν χάρη στην εμπειρία τους και την ε, επαγγελματική να εξυπηρετήσουν την οικονομική ανάπτυξη ανάκαμψη της Ευρώπης και γι' αυτό πιστεύω πως ήταν σημαντικό να υπάρχει να υπάρξει ένα δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο να μπορεί να θέσει στην διάθεση των επιχειρήσεων τη γνώση, την τεχνογνωσία αυτών των ε, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων πολιτών. Άλλη ιδέα έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες που δημιουργούν πλούτο σε τοπικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι επενδύσεις εγκύτητας είναι αυτές που πολύ συχνά επιλύουν ε, σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Η ιδέα ότι τα μεγάλα δημόσια έργα μπορούν να αποτελέσουν τη βασικό κινητήριο δύναμη για να βγούμε από την κρίση μπορεί να είναι απατηλή. Ε, θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα αντίβαρο σε σχέση με τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Μπορεί να λειτουργήσει ω μοχλό εξόδου από την κρίση, αλλά θα πρέπει να δοθεί εξίσου σημασία στι τοπικέ ε, επενδύσει που δημιουργούν τοπικά πλούτο. Έχουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο αυτέ οι επιχειρήσει και για να δημιουργηθεί πλούτο σε τοπικό επίπεδο και θέσει απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, καθώς και όλα τα θετικά, οι θετικές επιπτώσεις για την κοινότητα και για τις λιγότερο αστικές περιοχές είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισμός των ε, οικονομικών μέσων και φορολογικών κινήτρων ε, ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Είναι ίσως ε, δύσκολο το στίχημα, αλλά στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά για την αύξηση του ε, χώριου ακαθόριστου προϊόντος. Να, να παροτρινθεί η παραγωγικότητα μέσω από αυτό που εγώ αποκαλώ μία μικρομεσαία σημαίνει μία θέση εργασίας. Έχουμε 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάθε μία από αυτές θα δημιουργήσει μία θέση απασχόλησης έχουμε επιπλέον 20 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Πράγμα που θα ήταν τεράστια, ε, τεράστιο μέτρο και θα είχε μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Άλλη πτυχή των μικρομεσαίων έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε τη νέα εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δώσουμε ορατότητα και πεδίο δράσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Το έγγραφό μου δεν μπορούσε φυσικά παρά να αναφερθεί, όπως άλλωστε αναφέρεται και στον τίτλο, πως η καινοτομία είναι πολύ σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι είναι ένας πολύ σημαντικό κίνητρο για την ε, έξοδο από την κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να υπάρξει νέα εταιρική σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό κόσμο, ώστε να ωφεληθούν αμφότεροι. στήριξη στην ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί εξαρτάται το μέλλον της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και δύο πολύ σημαντικούς τομείς καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που πρόσφατα γνώρισε μεγάλη ύφεση και τέλος ε, την καινοτομία ώστε η βιομηχανία να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης σε αυτό το έγγραφο δεν μπορούσε να λείπει το σύστημα το εκπαιδευτικό, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στην αναζήτηση, στις θέσεις απασχόλησης, στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν νέες δεξιότητες, νέες ικανότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Ήδη μιλήσαμε για την δημογραφική πρόκληση. Για... Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν πάνω από 500 ε, εκατομμύρια ανθρώπων που ξεπερνούν ε, τα 60 χρόνια και ότι ξεπερνούν τον, τον αριθμό των ανθρώπων των παιδιών που, έχουν, που είναι άνω των 5 ετών. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και πρέπει να υπάρξει ένα αντίβαρο, δηλαδή η δραστήρια, η ενεργή γύρανση στην Ευρώπη από τη μια πλευρά και από την άλλη η διευκόλυνση των νέων για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ευρωπαϊκή οικονομία έχει να αντιμετωπίσει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους και γι' αυτό και ε, αυτή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που τίθενται σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και που εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να υπερασπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για, που συμβάλλουν στην συνοχή, όπως επίσης το ίδιο κάνουν και οι τοπικές ε, και οι, περι, οι γεωργικές ε, περιοχές. Σε όλα, ολόκληρη την Ευρώπη βλέπουμε απερίμωση των περιοχών της υπαίθρου με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις. Ε, που κάτι τέτοιο επιφέρει, ιδιαίτερα στο θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού και τα προβλήματα που σχετίζονται με την φτώχεια. Οι μικρομεσαίες αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό της αναζωγόνησης των ε, γεωργικών και τοπικών ε, ζωνών και επίσης είναι ένα σημαντικό μέσο κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. βιώσιμη ανάπτυξη ε, που θα πρέπει φυσικά να γίνει χρησιμοποιώντας πλήρως το δυναμικό της ε, κοινωνίας της ε, πληροφορίας με την εμπλοκή των τοπικών πληθυσμών στην ανάπτυξη και στην βιώσιμη ανάπτυξη κυρίως. Κλείνοντας, η ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Ζούμε μια εποχή πολύ δύσκολη και σοβαρή, εποχή προβληματισμού και λήψης πολιτικών αποφάσεων που θα είναι κρίσιμες ώστε να καθοριστεί το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Γνωρίζουμε ως ε, δίδαγμα από αυτή την κρίση ότι είναι απαραίτητο περισσότερο συντονισμός, εποπτεία και δέσμευση των ε, κρατών μελών ώστε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο να βρει σύμφωνες και τις επόμενες γενναίες. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τη φιλοδοξία για να έχουμε μια Ευρώπη που να βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο, που να μπορεί να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, και που είναι πολιτικής και οικονομικής φύσης. Και θα έλεγα τέλος πως το ευρωπαϊκό σχέδιο, το, το ευρωπαϊκό όραμα ανέκαθεν ε, προχώρησε χάρη στην μεγάλη δυνατή βούληση των ηγετών του και Ελπίζω ότι οι σημερινοί ηγέτες θα μπορέσουν να δώσουν το απαραίτητο ρυθμό, την απαραίτητη δύναμη, όθηση ώστε οι πολιτικές αυτές να υλοποιηθούν και να έχουμε συνείδηση πως εδώ, σε αυτό το επίπεδο, το κοινοτικό, διακυβεύεται το ευρωπαϊκό όραμα. Σας ευχαριστώ, <clears throat> κυρία Μπάστος, για την εισαγωγή στο θέμα. Ας ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια, δηλαδή, κυρία Μπερές, και μετά θα ακούσουμε με τη σειρά τους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, που τροποποίησατε το χρονοδιάγραμμά μας ε, και το πρόγραμμα όπως το είχαμε φτιάξει αρχικά, διότι μπορούμε έτσι να έχουμε όλους τους εισηγητές, τους θεματικούς δηλαδή, πριν ολοκληρωθεί η έκθεση. Με τη Ρετζίνα Μπάστος κάναμε λίγες ζαβολιές ε, ως προς την προθεσμία. Είχαμε όμως την ευκαιρία ε, επικοινωνίας και προφορικής και γραπτής για να μας διαβιβάσει τις ε, ιδέες της. αυτό ήταν πραγματικά το ζήτημα στο συγκεκριμένο έγγραφο να Ε, δούμε αυτό το ζήτημα γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο και με ένα κριτικό βλέμμα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Μία όμως που είναι στην καρδιά όλων των ανησυχιών και των φροντίδων είναι η απασχόληση. Οι μεγάλες εταιρείες αλλά και οι μικρές και οι μεσαίες κάνουν στρατηγικές για την τις εξαγωγές τους και εμεί θέλουμε να είναι δυναμικές και έχουν παρουσία εκτός των τυχών, αλλά γνωρίζουμε ότι σήμερα ε, οι μικρές εταιρείες, οι μικρές επιχειρήσεις είναι τα κοιτάσματα ε, ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και γι' αυτό θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Αυτό που είπατε για την ενιαία θηρίδα το σημειώνω και μου αρέσει πολύ, όπως επίσης και η ελληνική μεταξύ των γενεών, με την κινητοποίηση των παλαιότερων εργαζομένων, ε, των πρεσβυτέρων. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Και νομίζω και στην κοινωνία κινείται κάτι. Ανησυχούν βέβαια οι ηλικιωμένοι, αλλά Όλοι έχουν παιδιά και εγγόνια και καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν δυσκολίες και στις επόμενες γενιές και στις γενιές που θα αφήσουν πίσω τους. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να τους βοηθήσουν με εθελοντικό τρόπο και να δώσουν τη γνώση του τη σοφία του για να μειωθεί το βάρος που σηκώνει στους ώμου της η νεότερη γενιά, οι νεότερε γενιέ. Αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό και είναι καλό να κινητοποιούμε τη γνώση, την εμπειρία των ε, πιο ηλικιωμένων με τρόπο εθελοντικό για να συμμετέχουν εκεί και να διοργανώνουμε την αλληλεγγύη και μεταξύ των γενεών. Πολύ καλή ιδέα. Και ενδιαφέρουσα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρεται μερικά στοιχεία, τρία συγκρατώ. Το θέμα της κατάρτισης. Θα πρέπει να το δούμε αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή. Και από την αρχή έχουμε την ίδια δυσκολία σε δύο άλλα θέματα, που είναι ο κοινωνικός διάλογος, η οργάνωσή του ε, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η εξωτερική και εξωτερική ανάθεση κάποιων υπηρεσιών. Ακριβώ επειδή είναι μικρομεσαίε οι επιχειρήσει, αυτά τα τρία δεν μπορούν να τα υπομισθούν στο εσωτερικό τη εταιρεία και μπορεί κάποιο να τους βοηθήσει απ' έξω με πραγματογνωμοσύνη, γι' αυτό λέμε να δημιουργηθούν κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, ε, κατάρτισης με αμοιβαία ε, συμμετοχή και στον κοινωνικό διάλογο. Ε, δεν εννοώ εδώ κατακαιρματισμό ή δημιουργία ξεχωριστών δικαιωμάτων, ε, αλλά μια συλλογική προσπάθεια. Euh, και αυτά όλα πώς ε, κοστολογούνται. Γιατί αν μια μικρομεσαία επιχείρηση αναθέτει εξωτερικά κάποιες υπηρεσίες, δεν μπορεί να το κάνει με κόστος απεριόριστο, ας πούμε το λογιστήριο ή, τα συνεργεία καθαρισμού μπορεί να είναι εξωτερικά, να μην είναι της εταιρεία, αλλά κάπου να υπάρχει μια ε, λογική κόστους. Εναπόκειται στους υπόλοιπους συζητητές να δώσουν και εκείνοι τις ιδέες τους. Ε, ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Α, ακόμα συγγνώμη κάτι για την κατάρτιση λοιπον ε, πώς να το πω. Έχουμε κάποιες μεγάλες στρατηγικές φιλοδοξίες. Φερρυπίν στο περιβάλλον. Πολύ συγκεκριμένο αυτό το παράδειγμα. Και ξέρουμε και τι διακυβεύεται εκεί. Στο περιβάλλον, αν θεωρήσουμε ότι σημαίνει μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, δίκτυο διανομής κλπ. σε τοπικό επίπεδο, στην άλλη άκρη της οικονομικής αλυσίδας, αυτό μπορεί να σημαίνει ανανέωση των κατοικιών, βελτίωση των δημοσίων συγκοινωνιών, για παράδειγμα. Λοιπόν, ανανέωση ή ανακαίνιση των σπιτιών, αν πάμε μέχρι το τοπικό επίπεδο, τι θέλουμε εκεί, να έχουμε τεχνίτες εξειδικευμένους, ε, ωραίες μεγάλες φιλοδοξίες και τα μεγάλα σχέδια στις Βρυξέλλες. Αλλά επιτόπου ο τεχνίτης έχει την απαραίτητη ε, εκπαίδευση να ξέρει τι υλικά χρειάζονται για να είναι φιλικό προς το περιβάλλον το σπίτι, ο τρόπος που θα το ανακαινήσει. Και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό το Small Business Act και πώς αναθεωρείται. Γιατί το είχαμε δει και από την προηγούμενη θητεία. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Μπονσινιόρε. Θέλω να συγχαρώ την ε, συνάδελφο για την συμβολή που έκανε στις εργασίες μας. <clears throat> Να πω αμέσως ότι συμμερίζομαι τόσο. είπε και τις τελικές συστάσεις. το να θέσουμε στο επίκεντρο των ενεργειών μας ε, της μικρομεσίας είναι μια ενέργεια μεγάλη ευθύνης. Εμείς μπορεί να ευημερίσουμε μόνο αν μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Η φράση που λέει ότι η αναζήτηση του κέρδους θα πρέπει να συνοδεύεται από μεγάλη αίσθηση ευθύνης είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει κέρδος εάν δεν ε, δημιουργείται ταυτόχρονα θέσεις εργασίας. Εγώ πιστεύω πως καλύτερα είναι να ασχοληθούμε με το θέμα της βιώσιμης ευημερίας. Νομίζω πως είναι η ώρα να αρχίσουμε να λέμε ξεκάθαρα ότι στη Δύση ζούμε πάνω από τις πραγματικές μας δυνατότητες. Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε να πιστεύουμε την ανάπτυξη, ότι η ανάπτυξη θα συνεχίζεται με βάση τα χρέη. Πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας πλέον. Θα, Πρέπει να καταφέρουμε να εξηγήσουμε στις 27 χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ήρθε η ώρα να εξετάσουμε με ρεαλισμό την κατάστασή μας. Άρα λοιπόν η έννοια της ευημερία ε, πρέπει να εξηγηθεί καλύτερα. Δηλαδή ότι η εμφανή μας ευημερία είναι πάνω από τις δυνατότητές μας και ότι απαραίτητος πρέπει να αναπτυχθούμε περισσότερο αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα σημερινά επίπεδα ευημερίας. Και για να αναπτυχθούμε περισσότερο χρειάζεται μια θαραλέα πολιτική, ε, πολιτική που θα πρέπει πρώτη στον κόσμο να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω πως αυτές τις εργασίες θα ε, προκύψει μια τέτοιο είδους συμβολή. συμβολή. Και πάλι ευχαριστώ τη συνάδελφο που συνέταξε την έκθεση. Grazie Presidente. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο Μπάστος για την εξαίρετη της εργασία και κυρίως επειδή πολύ καλά περιέγραψε το ρόλο και τη σημασία του συστήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ιστορικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το πιο ευέλικτο κομμάτι της παραγωγικής δομής, τόσο της μεταποιητικής όσο και της, ε, των υπηρεσιών. Έχουν ε, δηλαδή παίξει πολλές φορές ε, το ρόλο του το ρόλο της αντικυκλικής λειτουργίας σε διάφορες φάσεις κρίσης από εκείνους περνά η δυνατότητα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και της διατήρησης σε πράγμα το οποίο ιδιαίτερα μου είναι σε εμένα, διατήρησης ε, το, σε παραγωγικής και μεταπητικής ε, και κτημένου της ε, Ευρώπης. Το να σκεφτεί κανείς ότι μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτή τη δομή στην Ευρώπη θα ήταν ανόητο και λαθασμένο. Και μόνο το προτείνει κανείς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αντίθετα, οι προτάσεις που μας κάνετε ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την αξιοποίηση αυτού του σημαντικού κομματιού του συστήματός μας. Για την αξιοποίηση πιστεύω πως είναι σημαντικό και εγώ να επιμείνουμε σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα. Το θέμα το οποίο εισάγει η Ρετζίνα, απλοποίηση δηλαδή της διοικητικών διαδικασιών, ισχύει για ολόκληρο το οικονομικό σύστημα στην ε, πράξη. Αλλά δεν διαφεύγει από κανέναν ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι για τις μεγάλες, γιατί τα διοικητικά κόστη ε, ή απλά και μόνο η αξία του χρόνου που χρησιμοποιείται για να λυθούν τα διοικητικά προβλήματα για τις μικρές επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Άρα λοιπόν η απλοποίηση είναι αυτή σημαντική αξία για όποιαδήποτε οικονομία και ακόμα περισσότερο για αυτούς που ε, για τους οποίους έχει μέσα στο πλαίσιο της δομής του κόστους, της λειτουργίας τους, μεγαλύτερο βάρος. Ενία θηρίδα, ναι. Δηλαδή, ολόκληρη αυτή η διαδικασία, ε, η οποία ε, πρέπει να γίνει σε διαφορετικό καμέρι για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, για την αλλαγή δραστηριότητας κτλ. Κάνει τις μικρομεσίες να χάνουν χρόνο αλλά και δημιουργεί συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Ενώ αν είναι μια ενιαία θηρίδα σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ε, πλήρης συντονισμός. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες από μόνες τους δεν μπορούν να το κάνουν, να μπουν σε μια θετική σχέση με το σύστημα που δημιουργεί ε, καινοτομία και γνώση. Τα πανεπιστήμια αλλά και μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις. Το κλειδί είναι να ε, παροτριθούν αυτές οι εταιρείε, επιχειρήσεις να λειτουργήσουν από κενού, σε συνεργασία. Στην αγορά μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά, αλλά όταν χρειάζονται καινοτομία και έρευνα, να μπορούν να πάνε μαζί στο χώρο που παράγει καινοτομία και έρευνα. Δηλαδή, το κίνητρο για να συνεργαστούν θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι για να γίνουν πολλά από αυτά τα πράγματα χρειάζεται μια θετική, ένα θετικό περιβάλλον. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικολογία εδώ. Μιλώ για το περιβάλλον γενικότερα, για το μέρος, ε, εκεί όπου γίνονται οι δραστηριότητες. Δηλαδή μια πόλη, μια περιφέρεια έχουν δυνητικά εντό του ε, τα στοιχεία για να βοηθήσουν με σημαντικό τρόπο την οικονομική ανάπτυξη και την ε, παραγωγική δραστηριότητα με προϋπόθεση ότι οι δομές τους θα είναι προς αυτό προσανατολισμένες. Γι' αυτό και πιστεύω Ε, θα πρέπει να δούμε τους τομείς. Ε, ορισμένες περιοχές ας πούμε ασχολούνται παραδοσιακά με το μετάξι, άλλοι με το μαλλί, άλλοι με τον ε, χάλιβα. Η αξία αυτή μπορεί να βοηθηθεί μέσω συγκεκριμένων στοχευμένων ενεργειών από πλευρά της διοίκησης. Δηλαδή, η δραστηριότητα της πόλης ή της περιφέρειας, ας πούμε, κατασκευή υποδομών, η ανάπτυξη κέντρων κατάρτιση είναι ένα σημαντικό μια σημαντική συμβολή στην αξιοποίηση της ε, ε, δαφικής ταυτότητας. Πολλές από τις επιχειρήσεις μας είναι πολύ σκορπισμένες και κάνουν λίγο απ' όλα σε πολλά μέρη, αλλά οι περισσότερες έχουν μια ταυτότητα περιφερειακή που για τις ίδιες αποτελεί ένα σήμα μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο πως πολύ συχνά η πρώτη ύλη συνδέεται και με το όνομα μιας πόλης ή με μιας περιφέρειας. Πιστεύω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρεται και στο έγγραφο της συναδέλφου Μπάστος, ίσως θα έπρεπε και να τον ισχύσουμε περισσότερο. Όλες μη των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου, ευχαριστώ και εκφράζω την εκτίμησή μου για την εργασία της κυρίας Μπάστος και βέβαια θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια ευρύτερη μεταποίηση στην Ευρώπη. Περισσότερο δηλαδή τη μεταποίηση εν τέλει. Και ασφαλώς αυτή που να βασιστεί στις προσπάθειες των μικρών και μεσών επιχειρήσεων, κανεί δεν το αμφισβητεί αυτό. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίζουμε επιχειρήσει οι οποίε δεν μπορούν να επιβιώσουν τι νόημα έχει να ναυπηγεί κανείς καράβια τα οποία κανείς δεν θέλει να αγοράσει. Είναι δαπανηρό, οδηγεί σε οικονομική καταστροφή. Ή επίσης όλα τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουμε. Κάποιοι αγοραστές πρέπει να βρεθούν για τα αυτοκίνητα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν σοφροσύνη όταν δαπανούμε τα χρήματα των φορολογουμένων ως κρατικές ενισχύσεις. Γενικό σχόλιο αυτό, φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Μερικά τώρα σύντομα σχόλια. Νομίζω ότι η έμφαση που δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σωστή και η πρόσβαση στην, σε πιστώσεις είναι σημαντική όπως είπατε. Να εξετάσουμε όμως και τι έγινε στις κεφαλαιαγορές όπου τα διάφορα επίπεδα απαιτήσεων για κεφάλαιο Παρ' όλα αυτά δεν εμπόδισαν τι ε, τράπεζε να φτάσουν σε ένα σημείο που να λένε ότι δεν έχουμε λεφτά πλέον για να δανείσουμε τι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει. Τώρα, η οδηγία περί υπηρεσιών είναι ουσιώδου σημασία για, να, για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη και για την παραγωγή πλούτου και ανάπτυξης. θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει κάνει πολύ καλύτερες προσπάθειες για να τα προωθήσει αυτά. Εξακολουθεί να μην υπάρχει, για παράδειγμα, η διακίνηση των ασθενών. Όλοι μας μεγαλώνουμε σε ηλικία. Και παρόλα αυτά η κινητικότητα δεν υπάρχει. Και ιδίω είναι κρίμα για εκείνους οι οποίοι δεν βρίσκουν κατάλληλες υπηρεσίες υγείας στις πατρίδες τους. Γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν τους ασθενείς αυτούς από το να διακινηθούν σε άλλες χώρες για να βρουν την υγειά τους. Για παράδειγμα, εμποδίζει την κίνηση αυτή σήμερα η Ισπανία. Ίσως μπορούμε να το πούμε αυτό καθαρά στην έκθεση τα συνταξιοδοτικά συστήματα επίσης. Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε βιώσιμα συνταξιοδοτικά συστήματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα σύστημα pay as you go, δηλαδή να βρίσκουμε ίσα ίσα τα χρήματα για να καλύπτουμε τις τρέχουσες δαπάνες. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα. Να δούμε και πότε θα παίρνουμε σύνταξη. Οι άνθρωποι γεννάνε όλο και περισσότερο μεταξύ 60 και 70 πρέπει να παίρνω σύνταξη. Μεταξύ 60 και 75 πρέπει να τα δούμε αυτά. Αυτά είναι σημαντικά και για τα δημόσια οικονομικά. Η παιδεία, οι ιδέες που περιλαμβάνει το κείμενο είναι καλές. Πολλοί λένε για 3% των εθνικών προπολογισμών για την παιδεία. Πολλές χώρες δεν το φτάνουν αυτό είπε ο Μπαρόσο ότι χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού MIT, Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Ένα e IT αυτή, η ιδέα όμως κάπου θαύτηκε σε κάποιο συρτάρι, σε κάποιο γραφειοκρατικό σιρτάρι της Κομισιόν, όμως εμένα η ιδέα αυτή μου είχε φανεί καλή. Γνωρίζω ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη που να μπορεί να ανταγωνιστεί το αμερικανικό MIT. Και δεν έχουμε τέτοιο πράγμα αλλά και τα διάφορα επίπεδα της παιδείας. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι εξετάσεις που λέγονται εξετάσεις πίζα. Τα βλέπει κανείς τα... τους μαθητές από 9 χρόνων μέχρι 18-19 βλέπουμε ότι όλο και μειώνονται οι αποδόσεις των μαθητών. Και τα λέω αυτά και στο γιο μου που μου λέει ότι δεν θέλω τόσο πολύ να μελετήσω, προτιμώ να ε, παίξω με τον υπολογιστή μου. Του τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί υπάρχουν για κάθε έναν Ευρωπαίο 5.000 φοιτητέ στην Ινδία ή στην Κίνα οι οποίοι δουλεύουν σκληρά και όταν θα μεγαλώσουν τα δικά μας τα παιδιά θα βρίσκουν δουλειά. Μιλήσατε και για την ευρωομάδα, την ομάδα του ευρώ και για συντονισμό των φορολογιών. Καλή ιδέα είναι και αυτή. Μήπω μπορείτε να μιλήσετε όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, γιατί αισθάνομαι σαν να με αποκλείεται διαρκώ. Μιλήσατε και για την EAS. Έχουμε μερικού εμπειρογνώμονε εδώ. Πώ θα λειτουργήσει αυτή, τέλο οι μελλοντικέ τάσει. Μιλείτε για τις δημογραφικές αλλαγές. Πραγματικά είναι ζωτική σημασία, αλλά νομίζω να προσθέσετε και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού που δεν την έχουμε. Δεν έχουμε κινητικότητα όπως θα μπορούσαμε να έχουμε. Τώρα η μετανάστευση. Χρειαζόμαστε τη, χρειαζόμαστε τη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε να έρθουν άνθρωποι εδώ και νομίζω ότι είναι καταστροφή αυτό που κάνουμε που προσπαθούμε να του διώξουμε. Ενώ σε λίγα χρόνια θα του πούμε ελάτε εδώ να δουλέψετε στην Ευρώπη και να φροντίσετε τους Ευρωπαίους που γυρνάνε. Το τελικό μου σχόλιο είπατε ή μάλλον λέτε εδώ στο κείμενό σας κάτι για παγκόσμιο αλλά τι εννοείτε λέτε να ληφθούν αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό που είχα μάθει εγώ Think globally, act locally να σκέφτεστε σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά να δράτε σε τοπικό ή εννοείται κάτι διαφορετικό που ε, θέλουν οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι απήχηση έχουν αποφάσει που λαμβάνουν και σε τοπικό επίπεδο. Αλλά ίσως μπορείτε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι εννοείται. Κλίντς. Γκίγκολτ. Χουντής, και Συγγνώμη συνάδελφοι, θα πρέπει να φύγω σύντομα, πολύ σύντομα κάποια σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ για το τόσο ενδιαφέρον έγγραφο, κυρίως για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μόνο κάποια συμπληρωματικά σχόλια που θα ήταν ενδιαφέροντα και για την έκθεση την ίδια. Αλλά δεν με ακούει η συγγήτρια. Μπο, δεν πειράζει. Βουαλά που λένε και οι Γάλλοι. Ναι. Α, εντάξει, τώρα ακούει. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω και να συμπληρωθεί στο έγγραφο είναι το εξής. Υπάρχει ένας μεγάλος κλάδος της οικονομία που τίνουμε να παραγνωρίζουμε ε, και να παραβλέπουμε το 10% του συνόλου της απασχόλησης δεν είναι ούτε στο δημόσιο τομέα, ούτε στον κλασικό ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, τις κλασικές εταιρείες που εντάσσονται σε συστήματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει ο λεγόμενος πλέον τρίτος τομέας, που δεν είναι ο τρίτογενής, προσέξτε, αλλά είναι η κοινωνική λεγόμενη οικονομία. Και θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε ε, και τι ειδικέ ανάγκες έχουμε εκεί και ποιες είναι οι ε, περιφερειακές αναπτυξιακές δυνατότητες. Σε αυτή την ε, προσπάθεια είναι πολύ φυσικός εταίρος. Ε, όταν θέλουμε να αναζωογονηθούν κάποιες περιφέρειες ή να διατηρηθεί η να διατηρηθει δραστηριότητα σε περιφέρειες της υπαίθρου, όπως το είπατε εσείς, ε, είναι σε δυσκολία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εμπειρία ε, και η γνώση αυτού του τρίτου τομέα της κοινωνικής οικονομίας για να διατηρείται η ε, ζωή σε αυτές τις περιφέρειες και στην Ήπεθρο. Μπορούμε λοιπόν να δανειστούμε μερικές από τις προτάσεις της έκθεσης Τόγια της περσινής χρονιάς που με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε στο Κοινοβούλιο για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκείνες που έχουν και πολλές κοινέ ανάγκες αλλά και πολλές ειδικέ ανάγκες διαφορετικές από εκείνες των άλλων. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή για να το προωθήσουμε. Κάτι άλλο. Αναζωογόνηση ε, της πολιτικής ανταγωνισμού. Θα βοηθούσε για να δώσει περισσότερο χώρο και στις μικρομεσαίες. Γιατί, από την άλλη, όλοι και περισσότερο βλέπουμε ε, ολιγοπολιακή οργάνωση των αγορών ε, και αυτό είναι απειλή. Και τέλος, νομίζω πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε κάποιες συστάσεις. Καλούμε γενικά για περισσότερα φορολογικά κίνητρα. Εγώ ως πρόσωπο ε, συχνά είμαι πολύ επιφυλακτικός για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα ε, κίνητρα, γιατί περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετές επιπλοκές και προβλήματα ε, στη φορολογία. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε και άλλο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός αυτών, πάντως, γενικά συμφωνώ ε, με τη γραμμή της συζητήτριας και τον κορμό της και τα γνωρίζει και η ίδια. Και βέβαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα μόνο τμήμα του τίτλου ε, του εγγράφου εργασίας και τώρα δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε ε, τα θέματα, τα νομισματικά και τα χρηματοοικονομικά για τη στρατηγική εξόδο από την κρίση και για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό νομίζω είχε ήδη καλυφθεί από προηγούμενα έγγραφα. Αυτά. Νομίζω θα επανέλθετε στα θέματα αυτά εσείς για να μην χαθούν οι ιδέες μας στην τελική έκθεση και προσβλέπω πάρα πολύ σε μεγάλη προσέλευση, να είναι γεμάτη η αίθουσα όταν θα συζητάμε την έκθεσή σας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει και εγώ να φύγω τώρα. Κύριος Χουντής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για το κείμενο που μας κατέθεσε και για τις σκέψεις που έχει διατυπώσει προκειμένου να συμβάλλει στην όλη προσπάθεια που κάνουμε. Θα ήθελα να πω ότι μιας και αρχίζουμε και τη μαζεύουμε τη συζήτηση, δηλαδή με το κείμενο της εισηγήτριας της Γενικής και τη συμβολή όλων, ε, θα ήθελα με αφορμή το κείμενο της ε, εισηγήτριας το σημερινό να πω ορισμένε και διαφωνίες μου, θα έλεγα και ερωτήσεις, μιας και σε βασικά θέματα της έκθεσης της εισηγήτριας δεν συμφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη συζήτηση που έχουμε κάνει. Επομένως, δεν είναι ακριβώς για το κείμενο, αλλά είναι σε ορισμένα βασικές διαπιστώσεις που κάνει το κείμενο. Και ε, συμφωνώ με τη σημασία που έχουν οι μικρέ μικρές, και, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη για την ανάπτυξη, στην τοποθέτηση του ζητήματος. Υπάρχει βεβαίως για μένα ένα ερωτηματικό τι εννοούμε μικρή και μεσαία επιχείρηση μέχρι που φτάνει ε, με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων, του επενδυμένου κεφαλαίου, αλλά πάση περιπτώσει α πούμε ότι το βρίσκουμε αυτό τι εννοούμε. Γιατί πολλές φορές είναι διάκριτο. Η πρώτη παρατήρηση είναι από πού η εισηγήτρια θεωρεί ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ένωσης. Το ερώτημα είναι τι είναι αυτή η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αν είναι υπολείμματα του παλιού κοινωνικού κράτους για το οποίο ήταν υπερήφανη η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, φοβάμαι πως μιλάμε για υπολείμματα αυτού του κοινωνικού κράτους. Αν μιλάμε στη λογική ότι έχουμε απελευθέρωση των αγορών, κριτήριο το κέρδος και εξ υπολείπου ασκείται κοινωνική πολιτική, νομίζω τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, τίθεται ένα ερώτημα. Θεωρούμε ότι είναι επίτευγμα της Ένωσης η κοινωνική οικονομία της αγοράς και μάλιστα αν κανείς κάνει την κοινωνική ακτινογραφία της Ευρώπης, 20 και πάνω εκατομμύρια άνεργοι, 50 ίσως και παραπάνω κάτω από το όριο της φτώχειας. Μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Το ερώτημα τίθεται πιο δραματικά θα έλεγα, τι ακριβώς είναι αυτή η κοινωνική οικονομία της αγοράς και για την οποία δεν ξέρω, φοβάμαι γιατί περηφανευόμαστε ότι είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Και το λέω αυτό διότι προφανώ είναι το νέο πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει και η μικρομεχαία επιχείρηση και άλλα ζητήματα. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπω τίθεται, και όχι μόνο σε αυτό το κοινωνικό το κείμενο, ο ανταγωνισμό κατανοείται ή παρουσιάζεται σαν μια ευγενή άμυλα μεταξύ μαθητών, τον, του γιου του κυρίου Σμιτ και άλλων, ποιο θα πάρει τον καλύτερο βαθμό στο σχολείο. Είναι μια ευγενή άμυλα. Αυτό είναι ο ανταγωνισμό κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό. Ε, είναι μια σκληρή, ένας πόλεμος μεταξύ των επιχειρήσεων για μεγαλύτερο κέρδος, να μειώσουν το εργασιακό κόστος, να πετύχουν μονοπωλιακές τιμές. Είναι μια άγρια κατάσταση. Μέσα σε αυτή την άγρια κατάσταση που τη βλέπουμε να εξελίσσεται, το ερώτημα τίθεται πώς μπορούν να επιβιώσουν απέναντι στις πολυεθνικές, χωρίς ιδιαίτερη προστασία, στις πολυεθνικές, αυτόν τον άγριο ανταγωνισμό, που στο τέλος βεβαίως καταλήγει σε συμπίωση του μισθού των εργαζομένων κτλ. κτλ πώς μπορούν να αντέξουν και ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντέξουν αν αφαιθούν και μάλιστα κατά την εισηγήτρια να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Αν είναι έτσι ο ανταγωνισμός δεν νομίζω ότι θα επιβιώσουν. Εδώ βεβαίω για να μην είμαι και εγώ επιπόλαιος θα ε, ε, είχε μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι η πορεία, θέλετε την τελευταία δεκαετία, αυτή τη δεκαετία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή πόσες υπάρχουν ακόμα, πόσες κλείνουν, πόσες ανοίγουν, ποια είναι η θέση τους. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε αν μπορούν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια και κατά την άποψή μου, και δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη γνώμη τουλάχιστον εδώ, ότι ο ανταγωνισμό δεν είναι ε, ροδοπέταλα, αλλά είναι μια σκληρή μάχη μεταξύ των επιχειρήσεων και οι κυρίαρχε, ε, το αναφέρθηκε και ο προηγούμενο ε, ομιλητή, έχουμε δεσπόζουσε θέσει, έχουμε μονοπωλιακέ καταστάσει που δεν αφήνουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να επιβιώσουν. Πιο σύντομα τώρα, γιατί είναι κάπω επιμέρου. Έχω ένα ερωτηματικό. Καλή ακούγεται αυτή η ιδέα για τους βετεράνους. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει. Το να παρατείνουμε τον εργασιακό βίο και το έχουμε συζητήσει μέχρι πού. Στο όνομα μιας εμπειρίας. Πράγματι υπάρχει εμπειρία. Αλλά αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να μεταβιβάζεται από τους εργαζόμενους τους νεότερους καθώς ας πούμε ανανεώνεται η θέση εργασίας κτλ. Δεν το καταλαβαίνω το σχήμα. Ακούγεται μια καλή ιδέα, δεν κατάλαβα το σχήμα. Αν όμως αυτό αξιοποιείται για να μεγαλώσει ο εργάσιμος βίος, δεν το βλέπω ότι είναι μια πρόταση, εν πάση περιπτώσει, που φέρνει σχετική κάποια ευημερία ή βελτιώνει τις συνθήκες ζωής. Τρίτη, ε, δεύτερη επιμέρους παρατήρηση και αυτή ξέρω ότι είναι αντικείμενο μεγάλου διαλόγου. Εμένα να σας πω κύριε συνάδελφοι, όταν ακούω σύνδεση της παιδείας, της εκπαίδευσης με την αγορά, ανησυχώ πάρα πολύ. Ανησυχώ πάρα πολύ διότι αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της παιδείας, της μόρφωση και περιορισμού του περιεχόμενου, του πανεπιστημιακού περιεχόμενου που πρέπει να έχει παιδεία. Το βλέπω στη χώρα μου, το βλέπω σε αρκετέ χώρε. Αν η παιδεία είναι εργαλείο για τις επιχειρήσεις και για την οικονομία απλώς και δεν, έχει, δεν είναι αυταξία, τότε νομίζω ότι πάμε πολύ πίσω από τις δημοκρατικές, πολιτιστικέ, ιστορικέ παραδόσει τη Ευρώπη. Το φοβάμαι, σα το καταθέτω και επομένω επιφυλακτικά ακούω αυτέ τι ε, τοποθετήσει. Δεν θα φάω περισσότερο χρόνο λέγοντας ότι για μια σειρά ζητήματα που ίσως ε, και το δικό μου χαρτί είχε αναφέρει πώς το βλέπουμε το δημογραφικό και το ασφαλιστικό και θα καταλήξω ότι προφανώς ανάμεσα στα άλλα αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση τα λέει κανείς και όχι μόνο εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν θα πάρουν λεφτά οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις από τα πακέτα στήριξης των κυβερνήσεων διατυπώνεται μονίμως το παράπονο ότι δεν πήγαν προς τις τράπεζες, δεν πήγαν στην πραγματική οικονομία, δεν πήγαν στις μικρές επιχειρήσεις. Επομένως, πέραν των άλλων, έχω ξαναδιατυπώσει αυτή την ιδέα, πιθανόν μέσα σε μια αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος να βοηθάει η ίδρυση τραπεζών ειδικού, ειδικού σκοπού, τράπεζες που να χρηματοδοτούν κατά προτεραιότητα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατόπιν τούτου και βεβαίως θα τα πούμε συνολικά, η δική μου διαφωνία είναι ριζική. Η εισηγήτρια τεκμηριωμένα και με την προσπάθεια που έκανε σημαίνει συνεχίζουμε το ίδιο παραγωγικό μοντέλο και ενισχύουμε την θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το ίδιο ευρωπαϊκό α το πούμε παραγωγικό μοντέλο. Η δική μου άποψη είναι ότι αν δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, δεν θα έχουν επιβίωση ούτε και μικρέ και μικρέ μεσαίε επιχειρήσει και δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται από τη μέχρι τώρα πορεία και ιδιαίτερα μέσα από τα συμπεράσματα τη κρίση. Ευχαριστώ. Donata Hübner. Thank you very much and I Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με την κοινωνική οικονομία της αγοράς, γιατί κανένα δεν το έχει πει μέχρι τώρα, ότι δηλαδή η κοινωνική οικονομία της αγοράς, ό,τι και να είναι, πάντως την γράφει η νέα συνθήκη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να την λάβουμε υπόψη. Και θα πω μάλιστα ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς μας έχει δώσει κάποια ανθεκτικότητα και μέσα στη χειρότερη φάση της κρίσης. Και η γνώμη μου είναι ότι και το βασικό στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που νομίζω ότι είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, απειλείται τώρα να καταστραφεί μέσα σε αυτήν την πολυσχηδή κρίση και η οποία είναι και τόσο πια μακροχρόνια και ε, έχει όπως είπα τόσες πτυχές που δεν μπορούμε καν να τις συλλάβουμε όλες ε, για την ώρα. Άρα πρέπει και να σκεφτούμε κιόλας ότι η ανοχή στην ανισότητα που ποτέ δεν ήταν τόσο υψηλή στην Ευρώπη όσο για παράδειγμα στις ΗΠΑ θα μειωθεί και άλλο στο μέλλον και ο κόσμος γίνεται πιο ευαίσθητος στο σχίσμα κοινωνικού εισοδήματο. και υπάρχει και ανοίγεται και ένα παράθυρο σε ένα νέο λαϊκισμό που κατά τη γνώμη μου θα περάσει σε όλες τις πολιτικές οικογένειες και θα μειωθεί, θα αποδυναμωθεί και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Διαβλέπω και ένα κίνδυνο να κάνουμε πολλές παραχωρήσεις, δημοσιονομικές παραχωρήσεις. Θα έχουμε το δίλημα δηλαδή να αυξήσουμε τις συντάξεις ή να δώσουμε περισσότερα λεφτά καλύτερα στην παιδεία, να δώσουμε τα λεφτά καλύτερα στην δημόσια έρευνα ή σε κρατικές ενισχύσεις για κάποιες υφιστάμενες βιομηχανίες οι οποίες εξακολουθούν ενδεχομένω να παράγουν απασχόληση. Στο μέλλον λοιπόν θα έχουμε και πολλές αντιφατικές δημοσιονομικές ανάγκες που ε, θα κάνουν βέβαια την, ε, τον εξισκελισμό των ε, προϋπολογισμών ακόμα δυσκολότερο από ό,τι είναι σήμερα. Και μάλιστα με ευκαιρία την έκθεση αυτή που μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες Νομίζω πρέπει να θέσουμε και το θέμα το θέμα της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς. Διότι αναμένουμε από τους δημόσιους θεσμούς, από τις κυβερνήσεις, να κάνουν πληθώρα πραγμάτων που δεν κατάφεραν να τα κάνουν και πριν από την κρίση. Και η καλή πολιτική υποτίθεται πρέπει να ασκείται για να δημιουργήσει ένα κλίμα ε, εφορίας, ένα κλίμα δηλαδή ε, κατάλληλο για να ανθίσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ποτέ θα ήταν και καθήκον των κυβερνήσεων και δεν έγινε. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε ε, ποιε είναι οι συνέπειες από, την, από το ότι η εμπιστοσύνη προς τους δημόσιου θεσμού και τις κυβερνήσεις θα εξαρτηθεί πολύ από την αποτελεσματικότητα αυτών των φορέων και από τη δυνατότητά τους να προσφέρουν και κοινωνικές υπηρεσίες ε, μακροπρόθεσμα. Και το πιο πιθανόν είναι, αν εξετάσετε τον ρόλο των κυβερνήσεων σήμερα και όλα αυτά τα πακέτα δημοσιονομικών κινήτρων, μπορεί να έχουμε δημόσιους φορείς στο μέλλον που θα μεγαλώσουν, που θα έχουν περισσότερα πράγματα να κάνουν, θα είναι περισσότερα και τα καθήκοντά τους από ότι μέχρι τώρα, από ότι πριν θα είναι επομένως και υψηλότερο το κόστος ε, για τον φορολογούμενο και δεν ξέρω αν αυτό είναι ιδεώδες για μας. Θα έχουμε λοιπόν ένα αυξανόμενο κόστο της κρατικής παρέμβασης και των κρατικών φορέων και μπορεί αυτό να οδηγήσει πάλι σε ε, αρνητική στάση απέναντι στις κυβερνήσεις και άρα να αποδυναμώσει την σταθερότητα των χωρών μελών. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα εξετάσουμε όταν μιλούμε για την ποιότητα της κρατικής παρέμβασης στα επόμενα χρόνια για τη δημιουργία πολιτικών που χρειαζόμαστε εν τέλει. Το δεύτερο θέμα που μου φαίνεται πολύ σημαντικό και που μου φαίνεται ότι οδηγεί την έκθεση ε, να συζητήσει αυτό το μεγάλο ρόλο της καινοτομίας είναι ότι η κρίση προκάλεσε τεράστια κενά στην παραγωγή. Και τώρα οι δημόσιες πολιτικές στοχεύουν περισσότερο στο να εξαλειφθούν αυτά τα κενά της παραγωγής. Η γνώμη μου είναι ότι δεν δίνουμε αρκετή σημασία στο κέρδος παραγωγικότητας, στην αύξηση παραγωγικότητας δηλαδή, που θα έπρεπε να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Να υπάρξει δηλαδή υψηλότερη παραγωγικότητα για να εξυπηρετήσει και τις κοινωνίες του μέλλοντος. Υποστηρίζω την έμφαση που δίνεται στην έκθεση στην καινοτομία και αυτό δεν θα σας εκπλήξει, διότι οι περισσότερες δουλειές, η περισσότερη απασχόληση θα προέλθει από καινοτόμε επιχειρήσεις με στραμμένα τα βλέμματα στο μέλλον, σε νέους τομείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω να το τονίσει κανένας. Νομίζω όμως ότι ε, εξετάζοντας τώρα τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξή τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα αντιμετωπίσουν στα επόμενα χρόνια, και νομίζω αυτό εννοούσε και ο Λεσμίτ, είναι αυτή η ιστορία της χρηματοδότησης των μικρομεσών επιχειρήσεων. Εάν θέλουμε καινοτόμε επιχειρήσει στο μέλλον, χρειαζόμαστε και πολύ risk capital. Χρειαζόμαστε δηλαδή χρηματοδότηση, η οποία να μπορεί να λάβει υπόψη και την υψηλή διακινδύνευση που έχουν οι υποθέσει αυτέ και χρειαζόμαστε και ένα είδος, ε, ε, ένα financial engineering που θα επιτρέψει στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να έχουν και πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Υπάρχει και ένας άλλος φραγμός που πρόκειψε στο πλαίσιο της Κοπενχάγης που η Κοπενχάγη εν τέλει δεν ήταν απόλυτη αποτυχία. Μιλάμε για οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα με, με χαμηλή δηλαδή εκπομπή διοξιδίων του άνθρακος. Αυτό δεν πρόκειται να το πετύχουμε εάν οι επιχειρήσεις δεν στραφούν σύντομα σε νέες, αν δεν έχουν δηλαδή νέες προδιαγραφές που να καλούνται να εφαρμόσουν για την παραγωγή. Οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις βρίσκονται σε σύγχυση. Δεν ξέρουν ακριβώς που πάμε. Μιλάμε για μείωση των διοξιδίων του άνθρακος κατά 20%, κατά 30%. Δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν είναι κατάλληλο για τις μικρέ και για επιχειρήσεις. Και το τελευταίο σχόλιο, πάλι ο Όλες το είπε, είναι η κινητικότητα. Τίνουμε να λησμονούμε ότι στην Ευρώπη η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, να μην πω ότι είναι μηδενική, αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Λόγω και του τρόπου που λειτουργεί η ενιαία αγορά, λόγω και του ότι η δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Υπάρχουν λοιπόν τόσα διαρθρωτικά ζητήματα που μπορούμε να βελτιώσουμε για να βελτιώσουμε έτσι και την ε, μοίρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μπαίνει και η κρίση στη μέση. Μπαίνουν πράγματα λοιπόν όμως που πρέπει να κάνουμε και που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε πριν από την κρίση. Η θέλει να τοποθετηθεί σύντομα και μετά... Α, προτιμάς το τέλος. Καλά, καλά λοιπόν ο Άλντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Μπάστος. Ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Μετά από όσα είπε η κυρία Μπάστος, ο Όλε Σμιτ το έθιξε η κυρία Χιούμπνερ επίσης, για την πρόσβαση στα κεφάλαια. Η κυρία Μπάστος είπε ότι είναι χρήσιμο να αρχίσουν να ρέουν οι πιστώσεις όχι οι πιστώσεις και οι αγορές των μετοχών, τα χρηματιστήρια, equities. Και τι συμβαίνει στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ευρώπη. Τα κεφάλαια, τα κερδοσκοπικά τώρα ακούμε ότι επιτίθενται στο ευρώ, επιτίθενται δεν ξέρω πού και τα ρίχνουμε στους κερδοσκόπους. Ε, εμείς οι πολιτικοί συχνά τίνουμε να το κάνουμε αυτό αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό, είναι λίγο άτοπο. Τι θέλει το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο θέλει να επενδύσει κάπου που να κερδίσει. Και όταν είναι τόσο πτυτική η οικονομία όσο είναι τώρα, ε, το κεφάλαιο κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, σπέκουλα είναι και κερδοσκοπία ε, και με τα νομίσματα και με τα κρατικά χρέη και με τις εταιρείε για να βγάλει γρήγορα κέρδος. Αυτό που θέλουμε εμείς όμως δεν είναι κεφάλαιο που να τρέχει ηλικιωδώς, αλλά ένα κεφάλαιο που να θέλει να παραμείνει ε, μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη. Και πώς λύνεται αυτό νομοθετικά. Είναι, πιστεύω εγώ, να εθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις και ε, τον ιδιωτικό τομέα και αυτό μπαίνει και ε, στα διαρθρωτικά ταμεία, να βάζουν κεφάλαια κινδύνου και να είναι ε, συμφέρον να επενδύουν εκεί σε μετοχές και με τις ΔΕΤ με συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αλλά με συγκεκριμένο στόχο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόμες, να είναι σωστά στημένο το σύστημα. Φανταστείτε ένα ποτήρι νερό που χύνεται στο τραπέζι. Εμείς τι κάνουμε σπίτι μας, παίρνουμε ένα σφουγγάρι και το μαζεύουμε. Ε, το ίδιο έγινε και εδώ, ακόμα και τεράστια οικονομική κρίση. Χύνεται, ξεχύνεται παντού το κεφάλαιο και ψάχνει ε, να βρει πού θα επενδυθεί. Εμείς χρειαζόμαστε ένα σφουγγάρι τώρα για να απορροφήσουμε αυτό το κεφάλαιο που υπάρχει, για να διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα εκεί που μας χρειάζονται, που είναι δηλαδή στις μικρομεσαίες θέλουν τα λεφτά να φέρουν και άλλα λεφτά, οι μικρομεσαίες θέλουν κεφάλαια. Ε, θα παντρέψουμε αυτά τα δύο. Γιατί ε, θέτουμε πολύ ε, το κέντρο βάρους στο χρέος. Έχει δίκιο ο κύριος Μποσσινιόρε που λέει ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Όντως. Και θα πρέπει βεβαίως να ε, πάμε στη χρηματοδότηση όχι μέσω χρέους αλλά μέσω επενδύσεων ενεργητικών. Κύριο κύριος Κλίντς, είχα γράψει και εγώ τον εαυτό μου στην ημερήσια, στον κατάλογο των ομιλητών και η κυρία Ροτμάιερ και τελευταία θα μιλήσει λίγο και θα συνοψίσει και η Περβάνς Μπερές και η κυρία Μπάστος. Σήμερα το πρωί ήμουνα σε ένα πάνελ, σε μια διάσκεψη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν αυτό ακριβώς που είπατε τώρα. Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια. Και επί της ουσίας θα πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι νέο το πρόβλημα. Και πριν από χρόνια υπήρχε αυτό ξανά και ξανά. Και ε, από παλιά και η πολιτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη-μέλη έκαναν μεγαλόστομες δηλώσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ραχοκοκαλιά της οικονομίας, θα σας στηρίξουμε και μια τρύπα στο νερό. Και το Small Business Act υπάρχει, αλλά τι γίνεται με την υλοποίηση. Ας τα αφήσουμε αυτό τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιούργησαν τις ε, θέσεις απασχόλησης, όλα αυτά τα εκατομμύρια θέσεων που είχαμε μέχρι την κρίση και μετά τις χάσαμε και είναι κρυφοί αφανείς πρωταθλητές, hidden champions τους λένε αυτούς ε, τους μικρομεσαίους. Λοιπόν, αν θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα κεφάλαια, το είπε και ο Άρτης προηγουμένως, στην Ευρώπη μόνο 30% παίρνουμε χρήματα από τις αγορές και 70% από τις τράπεζες. Στην Αμερική είναι αντίστροφα. Δεν λέω να γίνουμε Αμερική, αλλά δεν θα πρέπει ενδεχομένω να αναπτύξουμε ειδικά χρηματιστήρια για τους μικρομεσαίους. Για τους μικρομεσαίους χρηματιστήρια για να αντλούν κεφάλαιο, equity, σε σε όλα τα κράτη έχουμε αναπτυξιακές τράπεζες, πολλές φορές κρατικές. Και στη Γερμανία. Αυτή λέγεται Credit Anstalt, ε, τράπεζα ανασυγκρότησης. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός σύνδεσμος αυτών των αναπτυξιακών τραπεζών των κρατών μελών. Για να μπορούμε να στηρίζουμε ε, μία χώρα την άλλη. Όποιος έχει πρόβλημα δηλαδή να μην αρχίζει από το μηδέν, αλλά να υπάρχει ε, ένας τέτοιος σύνδεσμος, μία ένωση τραπεζών αναπτυξιακών όμως, ε, για να βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Εάν θέλει ε, μια εταιρεία μικρομεσαία να έχει δραστηριότητα διασυνοριακή, πρέπει στην άλλη χώρα να τρέχει να ψάχνει χρηματοδότηση από την τράπεζα από το μηδέν. Μετά, αν θέλει κάποιο να κάνει ένα δίπλωμα βρισιτεχνία, μία πατέντα, δεν μπορεί να τρέχει σε 27 χώρε να το κατοχυρώσει. Καταλαβαίνετε τι κοστίζει αυτό. Και ε, τυποποίηση ε, και κάποια εναρμόνιση. Α πούμε, μια μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε πέντε ε, κράτη να ξέρει πού κινείται και φορολογικά στις υπόλοιπες χώρες, όπως και στη χώρα του. Και να μην τρέχει να ψάχνει τους διάφορους συντελεστές που ισχύουν σε κάθε χώρα. Χρειάζεται λοιπόν και νοοτροπία ε, αλλαγή. Ε, Στι Ηνωμένε Πολιτείε σου λένε εντάξει, έχασε. Αλλά δεν πειράζει, α έχει και δεύτερη ευκαιρία. Ε, give a loser a second chance. Δηλαδή, αν κάποιο προσπαθεί ε, κάτι ε, να κάνει, μια καινοτομία και αποτυγχάνει, δεν θα πρέπει για πάντα, για όλη τη ζωή να έχει μπει σε τίποτα τράπεζες δεδομένων τύπου τη Ρεσία και να αγωνίζεται όλη του τη ζωή πώ θα φύγει από αυτή τη λίστα. Να έχει και δεύτερη ευκαιρία. Στη Γερμανία 17 με 20% ε, είναι μετοχικό, μετοχικό κεφάλαιο ε, στη χρηματοδότηση και με την οδηγία τώρα που προετοιμάζουμε ε, δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο τη ζωή των εταιριών. Δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι ασίδοντε οι επενδυτικέ δραστηριότητε και να τι αφήνουμε τελείω ανεξέλεκτε. Όχι. Αλλά να μην του δένουμε και τα χέρια ενώ εδώ τις ευλώσεις ανταγωνισμού. Γιατί αλλιώ θα χάσουμε και αυτά τα κεφάλαια και αυτή την πηγή κεφαλαίων και θα στερέψει και αυτή η πηγή. Και ακριβώς αυτή είναι η πηγή που ε, χρηματοδοτεί τους πιο καινοτόμους επιχειρηματίες. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ε, στους κανονισμούς ε, για την τήρηση λογαριασμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πάλι να μην υπερβάλλουμε. Μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση ενδεχομένω στην Ευρώπη, αλλά πάντα με όσο γίνεται πιο απλό τρόπο και μη γραφειοκρατικό. Και με χρήση αρχών που να είναι ε, προσαρμοσμένες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το θέμα του fair value ε, είναι μεγάλη επιβάρυνση, δεν είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μικρομεσαίων. Πολλά θέματα λοιπόν για τις μικρομεσαίες, ειδικά πρέπει να σκεφτούμε και να πιέσουμε, αυτή τη φορά να μην μείνουμε μόνο στα λόγια, αλλά να δώσουμε και σάρκα και οστά σε αυτά που λέμε. Και τώρα έχω λοιπόν την κυρία Χολμάγερ και μετά την Περβάος και την κυρία Ρεγκίνα Μπάστος. Ε, Αγαπητέ Πρόεδρε, το θέμα με έχει απασχολήσει αυτό των private equity των μετοχών. Υπάρχουν σίγουρα μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ε, ε, βρουν χρήματα με μέσω μετοχών. Βλέποντας βέβαια τι δυνατότητες ή τι διάθεση έχουν οι επιχειρήσεις αυτές να επενδύσουν σε περιοχές της υπαίθρου, θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ελάχιστη. Εγώ ε, προέρχομαι από μια περιοχή όπου είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Πρόκειται λοιπόν για ε, περιοχή πολύ κοντά στο, σιδηρό, τότε το πάλι ποτέ σιδηρό παραπέτασμα. Το ίδιο λοιπόν, τις ίδιες εμπειρίες ε, έχουν και οι Τσέχοι συνάδελφοι μου βέβαια. Λοιπόν, όσο και να ε, προσπαθήσουμε, δεν επενδύουν οι επιχειρήσεις εκεί. Σημαντικό λοιπόν είναι η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων, των μικρών και επιχειρήσεων στην λεγόμενη private equity να υπάρχει, αλλά να μην λησμονούμε και την ανάγκη να υπάρχουν προγράμματα προώθησης των περιοχών της υπαίθρου για να εξευρίσκεται δηλαδή κεφάλαιο έστω και αν είναι μέσω περιφερειακών τραπεζών που ίσως χρειάζεται βέβαια κάποια υποστήριξη από ειδικές τράπεζες όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και να μην λησμονήσουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελείται μοναχά από μητροπολιτικές ε, περιφέρειες, αλλά και από πάρα πολλές περιοχές της Υπέθρου, οι οποίες πλήττονται από μια ε, έντονη τάση να επενδύονται όλα τα χρήματα στα Μητροπολιτικά Κέντρα, αφήνοντας, απογυμνώνοντας έτσι τις επαρχίες, απογυμνώνοντας έτσι τις περιοχές της Υπέθρου από επενδύσεις, άρα από απασχόληση και άρα εν τέλει από κόσμο που μεταναστεύει πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα με όλα τα σχετικά προβλήματα κοινωνικά και άλλα. Ενώ παλαιότερα υπήρχαν πιο υγιείς ε, συνθήκες, πιο υγιείς δομές στην Ήπεθρο. Η private equity λοιπόν είναι σημαντικό, αλλά μέχρι τώρα αντιμετωπίζουν τους, τις περιοχές αυτές της, το, της υπαίθρου με μεγάλη δυσπιστία. Για παράδειγμα, ακίνητα και γήπεδα δεν εκτιμώνται στην πραγματική τους αξία. Μου γνωστοποιήθηκε μια ε, περίπτωση στην ε, τσεχική πλευρά, όπου ένα νεόδμητο κτίριο εκτιμήθηκε στο 20 μόλις της 100 της αξίας του. Και αυτό μόνο διότι ε, εφόσον αντιμετωπίσει συγκεκριμένη επιχείρηση που δανείζεται την περίπτωση πτώχευσης και πολιθεί το ακίνητο αυτό, λόγω του μικρού ενδιαφέροντος δεν πρόκειται παρά να ε, μπορέσει να πολιθεί μέχρι το 20% της αξίας του. Ας μην λησμονούμε λοιπόν τις περιοχές της υπαίθρου, ας τις φέρουμε πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί και αυτές εξαρτώνται πάρα πολύ από τη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επενδύσουν. Υπερβάμψω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Τρία θέματα. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι μια έννοια που μπήκε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην πραγματικότητα όμως, πώς να το πω, κατάλαβα τελικά ότι επιδέχεται πολλές ερμηνείες η έννοια αυτή. Και θα πρέπει να προσέξουμε τι θα γράψουμε εκεί και τι θα αποδώσουμε σε αυτή την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αν δεν είμαστε σαφείς στο τι εννοούμε, πώς το ερμηνεύουμε, ε, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, η θεωρητική εμπνευστέ της κοινωνικής ε, οικονομίας αγοράς, αν θέλετε να επιστρέψουμε στα κείμενα, πιστεύουν ότι ο καταναλωτής, ο πολίτης, ο οικονομικός δράστης θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για να είναι ένας καλός κοινωνικός εταίρος και φορέας για να λειτουργεί σωστά η αγορά. Αυτό εννοεί. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική ε, διάσταση που να εξισορροπεί την ισχύ της αγοράς. Έχω αποκομίσει και κάποιες ε, αφιβολίε πλέον ως προς την έννοια αυτή τη κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και ε, βαθύνοντας τη σκέψη μου, ε, έχω ξανασκεφτεί αυτή την ιδέα από τότε που μπήκε στο Σύνταγμα ακόμα και έχω οριμάσει λίγο στη σκέψη και νομίζω ότι λίγο έχει παλιώσει αυτή η ιδέα και να προσέξουμε πώς χρησιμοποιείται σήμερα. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το διακύβευμα δεν είναι μόνο ο φτωχός να γίνει ένας φορέας στην κοινωνία, ένας καλός καταναλωτής στην αγορά. Ο φτωχός είναι κάποιος που θέλει να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε παιδεία, σε υγεία, πριν καν απευθυνθεί στην αγορά για να είναι. Ε, Πώ είσαι λοιπόν ένα καλό υποκείμενο στην αγορά. Δεν είναι μόνο να είσαι καλός καταναλωτής. Και δεν ε, ασχολείται αυτή η ερώτηση με τα κοινωνικά στοιχεία. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο θεωρητικό αυτό που λέω. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο επεκτείνομαι ε, και είναι και σημαντικό όμως όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη έννοια. Εγώ προτιμώ να αναφέρουμε καλύτερα την ανάγκη κοινωνικής πολιτικής για να εξισορροπείται η εσωτερική αγορά. Γιατί δεν θέλω να αφήνουμε έτσι στην αρχική αφησημία την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Δεν αρκεί να είναι κάποιος καταναλωτής για να λειτουργεί σωστά σε μια αγορά. Είδαμε στην κρίση ότι δεν αρκεί αυτό για να δημιουργήσει την ισότητα στην οποία εμείς προσβλέπουμε στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Παρατήρηση δεύτερη για την κινητικότητα. Στα τελευταία δέκα χρόνια, μετά τη στρατηγική της Λισαβόνας δηλαδή, είχαμε μια αιμονή. Ο κόσμος να κινείται, να μετακινείται. Και γιατί, επειδή δεν είμαστε αρκετά κινητικοί όσο είπα, δεν λειτουργούσε σωστά η αγορά μας, η αγορά εργασίας. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Κάποιος το ανέθεσε, το είπε η ε, κινητικότητα, το ξέρουν αυτό οι ευρωβουλευτέ. όταν μετακινείς από τη μια ε, χώρα στην άλλη, τα, ε, τα επικοινωνούν τα χιούμπνερ αυτά, ε, έχεις προβλήματα με τις κοινωνικές σου εισφορές, με τη σύνταξη, τα δικαιώματα. ο κόσμο εντάξει να αλλάζει δουλειά, να τρέχει από εδώ και από εκεί, αλλά μην χάνει υπερβολικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, θεμελιωμένα. Αφήστε δε που ε, πιέσαμε πάρα πολύ τον κόσμο να αποκτήσει ιδιοκτησία, να αγοράσει ε, το σπίτι στο οποίο μένει και μετά τι θα κάνει. Και πού είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών. Ο κόσμος γερνάει. Ωραία. Οι νεότερες γενιές τι θα κάνουν. Θα πρέπει να είναι κατέρωθεν η αλληλεγγύη. Εγώ δεν ονειρεύομαι έναν κόσμο όπου όλοι οι ηλικιωμένοι ε, να είναι εγκαταλελειμμένοι, σταθμευμένοι σε οίκους ευγυρία και όλοι οι νέοι να έχουν μετακινηθεί κάπου αλλού για να βρουν δουλειά, γιατί εδώ δεν έχει. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι στόχος αυτός αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας. Κινηθείτε για να δουλέψει η αγορά. Όχι. Ε, μπορούμε να το σκεφτούμε και διαφορετικά. Και αν είμαστε και συνεκτικοί με τους στόχους μας έτσι και συνεπείς, ας πούμε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, δεν θα πρέπει όλο να τρέχει 300 χιλιόμετρα κάθε φορά να πάει να δει το συγγενή του, τη μάνα του, την οικογένειά του. Εντάξει μετακίνηση, αλλά να εργάζονται κοντά. Με συγκοινωνίες δημόσιες, σε κοντινέ αποστάσεις, όχι χιλιάδε χιλιόμετρα. Ε, να δούμε και αυτό το θέμα της ανάπτυξης ε, της Ευρώπης, αλλά η αγορά δεν περνάει μόνο από την κινητικότητα των εργαζομένων. Και αυτοί που πραγματικά αλλάζουν γρήγορα και μετακινούνται είναι πολύ φτωχοί και πολύ πλούσιοι. Ε, ε, η μεγάλη μεσαία κατηγορία παραμένει κάπως ε, εγκατεστημένη κάπου. Τώρα, στην έκθεση της Ρεζίνα Μπάστος έχουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι. Είναι η Ειδική Επιτροπή για την Χρηματοοικονομική Κρίση, την Κοινωνική και την πιστοτική. Και κάποιο ε, μίλησε για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις και την πρόσβασή τους ε, στα κεφάλαια, εκτός του, του τραπεζικού συγγνώμη, συστήματος. Αν θέλουμε και πάλι να είμαστε συνεπείς, ε, πρέπει να, να πούμε ότι χρειάζονται και τα δύο συστήματα για να χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες. Θυμάσαι τη Βασιλεία 2 τι έγινε. Ήταν ένα από τα αντικείμενα και τα διακυβεύματα της διαπραγμάτευσης δεν ξέρω αν έχετε τα στοιχεία, αλλά είναι πολύ ε, μικρή η δημοσιότητα για το πώς χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά οι τράπεζες, ποιες είναι οι εταιρείε, ε, τι γίνεται και ακούμε όλα αυτά που ακούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρη εγώ τώρα που επανακαθορίζουμε τους κανόνες για τις τράπεζες αυτό θα έχει αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσει και να το λάβουμε υπόψη μα ποιο αντίκτυπο θα έχει. Αλλιώς δεν είμαστε συνεπείς. Τώρα, πώς θα έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια οι μικρομεσαίες εκτός των τραπεζών. Και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί όταν κάνουμε εμείς τη μεγάλη ε, νομοθεσία μας ε, προσπέκτους, δεσπόζουσα ε, θέση, κατάχρηση στην αγορά, όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά και η ιδέα του να έχουμε χρηματιστήρια των μικρομεσαίων είναι τελείως εκτός λογικής μας. Είναι καινούριο. Ε, στην οδηγία προσπέκτους που αναθεωρείται, το είδαμε αυτό. Αν θα πρέπει μια μικρομεσαία να το εφαρμόσει αυτό, κάηκε. Αλλιώς ε, ε, θα ασχολείται μόνο με αυτό. Και θα γίνει εξειδικευμένος οργανισμός και δεν θα κάνει καμιά άλλη δουλειά. Λοιπόν, να έχουμε όλα αυτά υπόψη μας, διότι αλλά λέμε ότι είναι πολύ σημαντικέ οι μικρομεσαίες να έχουν όμω και χρηματοδότηση και πρόσβαση με όρους ευνοϊκούς. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Περβάνς Μπερές και όλους τους ε, συμμετέχοντες στη συζήτηση για αυτό το θεματικό έγγραφο. Τελικά αυτό το έγγραφο έδωσε την έμφαση που επιθυμούσαμε ε, στις, ε, στο light motif του, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως κινητήρια δύναμη στο γενικό οικονομικό πλαίσιο, νομίζω πως έτσι πρέπει να δούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, της Ευρώπης, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέσο, είναι η Ευρώπη εμπειρογνώμονας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό και θα μπορούσαν να παίξουν κρίσιμο ρόλο για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Και είναι επίσης ένα σημαντικό μέσο, ένα εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή παίζουν ένα ρόλο μικρομεσαίες ε, κοινωνικής ευθύνης που είναι ε, διαφοροποιητικός. Έχουν μια εγκύτητα με τις ε, τοπικές κοινότητες που είναι πολύ σημαντικότερος με τις σε σχέση με τις πολυεθνικές ή τις μεγάλες επιχειρήσεις και επίσης έχουν μια κοινοτική φιλοσοφία και οικονομική φιλοσοφία που τις οδηγεί σε ένα ρόλο πολύ πιο... ένα ρόλο κοινωνικοποίησης ας πούμε ε, για την κάθε περιοχή. Νομίζω πως αυτά προέκυψαν από τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων ότι όντως δηλαδή εξυπηρετούν την κοινωνική οικονομία της αγοράς που είναι η ευρωπαϊκή μας οικονομία. Προτείνουμε, προτείνω στην εισαγωγή μου, στην εισήγησή μου, τόσο στο έγγραφο όσο και στην προφορική μου εισήγηση, ότι οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής οικονομίας της ε, αγοράς στην Ευρώπη, δηλαδή ελευθερία, αλληλεγγύη και αυτές είναι οι βασικές αξίες που θα δώσουν ε, σάρκα και οστά στα προγράμματα. Τώρα, λιγότερο φιλοσοφικά ζητήματα και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είναι αυτή μια σύσταση που κάνουμε στην έκθεσή μας για το Small Business Act. Βασικά πέντε είναι τα σημεία. Πρώτον, τι είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι σημαντικό να ορίσουμε εκ νέου να τροποποιηθούν οι μηχανισμοί λειτουργίας και δημιουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και εδώ αναφέρομαι και στα όσα είπε και ο συνάδελφος Κομφεράτη να διευκολυνθούν ε, οι δραστηριότητες η κοινωνική διάσταση πρέπει να δοθεί επίσης στις μικρομεσαίες και Επίσης καινοτομία, σύνδεση με τον ακαδημαϊκό κόσμο, όπως αυτό αναφέρθηκε στο έγγραφο. Και έπειτα αυτό το Small Business Act θα πρέπει να το ξαναδούμε όσον αφορά την ε, κινητοποίηση, τα κίνητρα προς τις μικρομεσαίες και την πρόσβαση στις αγορές. Να μπορεί δηλαδή αυτός ο επιχειρηματικός κλάδος να έχει μια ιδιαίτερη, να τύχει μια μεγαλύτερη προσοχή για προσανατολισμό τους και ε, πρόσβαση στην αγορά. Έπειτα, αξιοποίηση των ε, περιφερειακών ταυτοτήτων. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα μέσο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ε, την, ταυτότητα αυτή είναι τα κοινοτικά ταμεία. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή όσον αφορά την ταυτότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των περιφερειών στις οποίες είναι τώρα. Εκεί δεν μπορώ βέβαια εγώ να εξαλείψω όλες τις αμφιβολίες, αλλά αυτό που είπατε τι είναι σε μια κοινή ε, προσπάθεια, σφαιρική προσπάθεια. Υπάρχουν αναδυόμενες οικονομίες οι οποίες ανταγωνίζονται με τη δικιά μας. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό επίσης τέρο την ΕΥΠΑ και άρα εμείς πρέπει να επιβιώσουμε και να επιβιώσουμε με φιλόδοξο τρόπο στο μέσο αυτού του κόσμου που μας ε, διαρκώς μας εγκαλεί. Δηλαδή να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιο κόσμο ανήκουμε και να λειτουργούμε έχοντας υπόψη μας όλα αυτά, ότι πρέπει να είμαστε δηλαδή πιο φιλόδοξοι. Και να γνωρίζουμε επίση ποιε είναι και ποια είμαστε δικά μα ευαίσθητα σημεία. Δηλαδή, σε επίπεδο επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση στις πιστώσεις. Ε, δεν είναι βέβαια το πιο σημαντικό θέμα που αφορά την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά γνωρίζουμε πως αυτή την περίοδο οι μικρομεσαίες επιβιώνουν και έχουν ένα ρόλο ισχυρό ως ένα βασικό μέσο ένα βασικό μέσο έξοδο από την κρίση και οφείλουν να έχουν πρόσβαση, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην, ε, στις πιστώσεις. Ε, είτε δηλαδή, όπως είπε η Μπερές, με το τραπεζικά, τραπεζικές επιστώσεις, δημόσιες πιστώσεις ή μια, ε, ένα μείγμα αυτών των δυο. Γιατί ήδη είδαμε ότι το να εξαρτάται κανείς ε, υπερβολικά από ένας μόνο σημείο είναι, πολύ επικίνδυνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όπως ανέφερε και ο πρόεδρος Κλίνς, η αγορά συμβάλλει κατά το 30% και οι τράπεζες κατά το 60%. Πολλές φορές αυτό δημιουργεί εξάρτηση από έναν μοναδικό φορέα σε αυτό το περίπλοκο παιχνίδι. Δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω περισσότερο σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν. Θα ήθελα μόνο να πω, για να ολοκληρώσω, ότι η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα των οικονομικών φορέων είναι εξαιρετικά σημαντική. Για να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο το οποίο ανέφερε η συνάδελφος Χούμπνερ, είναι σημαντικό όλοι οι φορείς να έχουν εμπιστοσύνη στους πολιτικούς τους υπευθύνου για τη λήψη των αποφάσεων. Χωρί αυτή την εμπιστοσύνη δεν υπάρχει βιωσιμότητα, δεν υπάρχει βεβαιότητα, δεν υπάρχει πρόοδο. Όλα αυτά εξαρτώνται, από όλα αυτά μάλλον εξαρτάται και η επιβίωσή μας, να υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας φορείς. Ε, ευχαριστώ. την θεματική ε, συντονίστρια και την εισηγήτρια κυρία Μπερές. Τώρα τελειώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση αλλά και όλο το πρόγραμμα εργασίας. <laughs> Η Περβάνς βέβαια έχει ολοκληρώσει ε, την προσωρινή της έκθεση που περνάει τώρα στην μετάφραση και στις 18 Μαΐου στο Στρασβούργο θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, δούμε την ε, έκθεση αυτή, θα την υποβάλει δηλαδή υπερβάνω επίσημα πια. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν στις 18 Μαΐου. Χαίρομαι που ήσασταν τόσο πολύ άριθμοι σήμερα ένα απόγευμα Πέμπτης. Ευχαριστώ και πάλι την ε, θεματική συντονίστρια και σας ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω όλους πάλι στο Στασβούργο.